έλαβε μέρος το πρωί στην 33η διακοινοβουλευτική ε, συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας και είχε εξαιρετική συζήτηση και με τους ομολόγους της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν στην εξομάλυνση και την διόρθωση των αποκλήσεων